Μας περνούμε λοιπόν σε αιτιολογήσει ψήφου. Προς ενημέρωσή σας, Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και 4 του κανονισμού η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στη συνεδρίασή της στις 26 Μαρτίου 2012 επαλήθευσε τις εξουσίες και πρότεινε ομόφωνα να επικυρωθεί εξουσία των συναδέλφων Πέτρη Σαρβάμα από την 1η Μαρτίου και της Ρεμπέκα Τέιλορ από τις 8 Μαρτίου και μετά σας προτείνω να, τα, ε, να εγκρίνουμε τις εντολές. Επομένως δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση και εγκρίνονται. Έχω λάβει επίσης από το ΕΛΚΑ, τους σοσιαλιστές, την ΑΛΔΕ, ε, να συμπεριληφθούν σε επιτροπές ε, και αντιπροσωπείες, στην Επιτροπή Δημοσιονομικής Ελέγχου του Περιπολισμού κ. Άβελ, ε, στη θέση του κ. Κοζανίνο. Στην Επιτροπή Αναφορών η κυρία Τέιλορ δεν είναι τακτικό μέλος πια. Στην αντιπροσωπεία της συνεργασίας